Dear colleagues, dear colleagues, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Ω συνήθω, είναι δύσκολο το απόγευμα να αρχίσουμε στην ώρα μα, αλλά έχουμε μόνο μία ώρα και 30 λεπτά για τη συζήτηση και έχουμε έναν εξέχοντα προσκεκλημένο, μία εξέχοντα προσκεκλημένη, την κυρία Χριστιανά Φιγέρας, διοικητική γραμματέα του UNFCCC, δηλαδή της, ε, συμφωνίας, της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Καταρχάς την ευχαριστώ λοιπόν που είναι εδώ μαζί μας για το διάλογο εν ώψη της διάσκεψης ε, στο Παρίσι. Είναι πολύ κατάλληλη στιγμή γιατί η Επιτροπή μας στις 21 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσει την έκθεσή της με τίτλο «Προς μια νέα διεθνή συμφωνία το Παρίσι» που θα είναι και εντολή για την 15 μελή αντιπροσωπεία μας στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του τμήματος υψηλού επίπεδου της COP21. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση που αποτελεί κλιματική αλλαγή, να κάνουμε τα αναγκαία βήματα για να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Η συμφωνία στο COP21 στο Παρίσι, με βάση ένα φιλόδοξο και νομικά δεσμευτικό κείμενο που να είναι ανάλογο με το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου ενώ θα επιτρέψει την δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν όλα τα αναγκαία για να περιορίσουμε τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με αυτούς τους στόχους ψήφισε να υλοποιήσουμε τους στόχους της Δευτέρας περίοδου δέσμευσης του πρωτοκόλου του Κιώτο, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε την αναγκαία νέα τεχνολογία για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανάλογα με, την, με βάση τη δημιουργία ενός πράσινου ταμείου για το κλίμα και με τη δέσμευσή μας να υπάρξει συμπληρωματική χρηματοδότηση 100 δις ε, το χρόνο, δολάρια, είπα, μέχρι το 2020. Κυρία Φιγκέρας, έχετε το λόγο. Είμαι σίγουρο ότι η Επιτροπή μας θα σας ακούσει, προσδοκεί να σας ε, ακούσει για την ε, πορεία προς την ε, διάσκεψη αυτή και για την εκπλήρωση των προσδοκιών επίτευξη συμφωνίας σε αυτή τη διάσκεψη στο Παρίσι τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση να τα ξαναπούμε. Είναι πάντα θαυμάσιο να είμαι εδώ και με χαρά βλέπω μερικούς παλιούς φίλους και μερικούς νέους φίλους. Σας ευχαριστώ για την στήριξη που έχετε όλοι δώσει για την επικύρωση της δεύτερης περίοδου δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Ελπίζω τα κράτη-μέλη που ακόμη δεν έχουν εθνικός επικυρώσει να το κάνουν σύντομα και καταλαβαίνετε ότι από πολιτική σκοπιάς η επιβεβαίωση, η επικύρωση ότι όλες οι χώρες θα λάβουν νομικά δεσμευτικές αποφάσεις και θα τις εφαρμόσουν είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε ακριβώς πριν από το Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωση από τα κράτη-μέλη τους ώστε όλοι να προσθεθείτε στο κατάλογο των χωρών που έχουν επικυρώσει. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω για το πώς πάει η διαδικασία. Τώρα δεν θα σας κουράσω με τρομερές λεπτομέρειες, αλλά ίσως θέλετε να ξέρετε πού ακριβώς είμαστε στη διαδικασία. Και μετά να μπω σε μερικά θέματα που νομίζω είναι κοινού ενδιαφέροντος για όλους μας, που είναι η φιλοδοξία. Πώς θα καθορίσουμε τις φιλοδοξίες που έχουμε για το Παρίσι, για τη διαδικασία. Σίγουρα θα χαρείτε που θα σας πω ότι η δουλειά που κάνουμε τώρα είναι η εκπόνηση του πρώτου κειμένου της, της πραγματικής, δηλαδή του κειμένου που θα πρέπει να υπογραφεί στο Παρίσι. Ορισμένοι εργαζόμασταν τέσσερα χρόνια για αυτό το κείμενο και όποιος ε, έχει κυλοπονήσει τέσσερα χρόνια αισθάνεται τώρα ότι κάτι έχει αρχίσει και βγαίνει και πιστεύω ότι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα έχει βγει ολοκληρωτικά διότι θα ανακοινωθεί στη φάση που βρίσκεται το κείμενο για τη συμφωνία στο Παρίσι μαζί με την απόφαση που θα το συνοδεύσει. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική διαδικασία αυτή στην οποία έχουμε εμπλακεί και θα εκπλαγείται από το βαθμό προόδου που θα αντιπροσωπεύει αυτό το κείμενο σε σχέση με το υπάρχον κείμενο. Λοιπόν, περιμένετε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για κάτι που νομίζω ότι θα σας χαροποιήσει. Κατόπιν ξέρετε ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω διαδικασία, θα έχουμε μια συνεδρία στον Οκτώβριο, μια pre-COP τον Νοέμβριο και μετά έχουμε την COP στο Παρίσι. Όπου θα εγκρίνουμε, θα εγκρίνουμε μια συμφωνία στο Παρίσι και αν όλα καλά, πάνε όλα πάνε καλά, μπορεί να γίνει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς πολύ φασαρία. Θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, το περιεχόμενο. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας. Πολλές λεπτομέρειες θα περιληφθούν σε αυτή τη συμφωνία για το Παρίσι. Παρά το ότι είναι σύντομο το κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να συνοψίσω ποιοι είναι οι στόχοι μας πώς θα υιοθετήσουμε φιλόδοξους στόχους. Υπάρχουν τρεις καθοριστικοί παράγοντες που θα μας επιτρέψουν σιγά σιγά με βάση τη φωνή του Παρισίου να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους. Ο πρώτος που είναι η βασική, η βάση είναι το σύνολο των συνεισφορών από όλες ε, τις ε, πηγές, από όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση που την ευχαριστώ Έχουμε 62 εθνικές επιτροπές για την ε, διάσκεψη. Περιμένουμε να έχουμε περισσότερες μέχρι το τέλος της προθεσμίας. Με τις εθνικές συμβολές που έχουμε ήδη είμαστε περίπου στο 70% των παγκοσμίων εκπομπών. Θα πάμε λίγο πάνω από το 70% μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όμως αυτό δεν είναι η κατάληξη των φιλοδοξιών μας, είναι απλώς το σημείο αφετηρίας. Η ελάχιστη προσπάθεια που μπορούν να δεσμευθούν ότι θα κάνουν οι χώρες. Με τις υπάρχουσες τεχνολογίες και με τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις. Αλλά με πολλές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την ομοθέσια. Και αυτό είναι μάλλον μια, ένα δυναμικό των εθνικών ε, συνεισφορών που θα βοηθήσει ακριβώς να υιοθετηθούν διάφορα νομοθετήματα που θα προωθήσουν τους στόχους μας. Αυτές οι εθνικές συμφωνίες οπωσδήποτε δεν θα φτάσουν στους έξι βαθμούς. Στους δύο βαθμούς, συγγνώμη. Εάν λοιπόν προσπαθούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς να έχουμε μια δεσμευτική ε, συμφωνία, χωρίς την σύμβαση πλαίσιο, θα είχαμε μέχρι το τέλος του αιώνα 4 με 5 βαθμούς θέρμανση, ενώ με αυτές τις συμβολές των INDC θα έχουμε 3 βαθμούς. INDC είναι οι προτινόμενες εθνικές συμβολές. Αυτά τα INDC δεν είναι μόνο το ελάχιστο όριο που είναι διαφορετικό από το να μην αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά πέρα από φιλόδοξα INDC Στόχος μας είναι η Συμφωνία του Παρισιού να μην είναι στατική, αλλά να πυροδοτήσει μία διαδικασία πολλαπλασιαστική, ούτω ώστε ε, με την πάροδο του χρόνου να γινόμαστε όλο και πιο φιλόδοξοι, να περνάμε σε όλο και πιο φιλόδοξους στόχους. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό της συμφωνίας αυτής. Κάθε 5 με 10 χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ε, θα γίνεται, αλλά κάθε τόσο κάποιες χώρες θα έρχονται, θα συζητούν πώς θα έχουν πάει με τα NDC τους και θα βλέπουν αν είναι δυνατόν να αυξήσουν τις προσπαθίες τους. Και το τρίτο τμήμα για να υιοθετήσουμε φιλόδοξους στόχους είναι να έχουμε ένα σαφώς καθορισμένο και θεσμοθετημένο από τη συμφωνία τελικό στόχο. Δεν μπαίνει ποτέ σε κάποιο όχημα, τουλάχιστον σε δημόσια συγκοινωνία, χωρί να ξέρει που θα σε πάει. Μόνο αν ξέρει το στόχο σου. Μπορείς να πεις σε ποια φάση της διαδικασίας είσαι, εάν τον προσεγγίζεις το στόχο ή αν ενδεχομένω απομακρύνεσαι. Η διαλογική και τη συμφωνία του Παρισίου. Τα INDC θα πρέπει να είναι ορόσημα, αλλά πρέπει να έχουμε και τελικό προορισμό, ούτως ώστε κάθε ορόσημο στο οποίο θα φτάνουμε στην πορεία να μας βοηθάει να δούμε τι μας μένει. Ο τελικός στόχος είναι κλιματική ουδετερότητα τουλάχιστον το δεύτερο τμήμα του αιώνα μας. Δηλαδή να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εκπομπών που είναι αναπόφευκτες και τη φυσική δυνατότητα απορρόφησης εκπομπών του πλανήτη. Αυτά τα τρία τμήματα για μένα είναι μία τριάδα για το πώς θα καθορίσουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν ήδη επιτευχθεί, σημαίνει ότι έχουμε ένα σχέδιό τους, πρέπει όμως να επιβεβαιωθούν αυτά τα σχέδιά τους και να κατοχυρωθούν μέσω συμφωνίας του Παρίσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Πολλή δουλειά έχουμε ακόμη μπροστά μας. Όλοι όσοι θέλουμε η συμφωνία στο Παρίσι να είναι όσο πιο φιλόδοξη γίνεται. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι οι φιλοδοξοί αυτοί στόχοι δεν μπορούν να γίνουν αυτομάτως αποδεκτοί από 195 χώρες στο Παρίσι χωρίς την υποστήριξη των αναπτυσσομένων χωρών. Γιατί αυτή η τριάδα στόχων για τις αναπτυσσομένες χώρες σημαίνει αλλαγή, ριζική αλλαγή, θεμερική αλλαγή οικονομικού μοντέλου το οποίο ισχύει εδώ και 100 χρόνια και παραπάνω. Και μιλάμε για χώρε που πρέπει να εξασφαλίσουν τροφή και στέγηση πάνω από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπου. Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά τι αναπτυσσόμενε χώρε, έξω και η οικονομική υποστήριξη, η οικονομική βοήθεια είναι ζωτικής σημασία για την προσεχή περίοδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οικονομική και τεχνική βοήθεια προ τι χώρε αυτέ, αποτελεί σημαντικό σημαντικότατο κομμάτι του παζλ αυτού. Και να σημειώσω ένα κατακλείδι όσον αφορά τους στόχους ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία μπροστά μας που δεν την είχαμε τα τελευταία έξι χρόνια να αναγνωρίσουμε επισήμω τον ρόλο και τη συμμετοχή, τη συνεισφορά των μη κρατικών φορέων τη τοπική αυτοδιοίκηση, των δήμων, των περιφερειών, ε, εταιριών, οργανισμών, οργανώσεων και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί μαζί προχωρούμε προς τα εμπρός επιθετικά και θετικά θα έλεγα για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος. Θα αναγνωρίσουμε λοιπόν τη συνεισφορά όλων αυτών στο Παρίσι και θα αρχίσουμε να δεχόμαστε και στοιχεία για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τη συνεισφορά τους η οποία επικαλύπτεται εν μέρη με τις κρατικές συνεισφορές αλλά σε κάθε περίπτωση βοηθάει τα κράτη-μέλη, τι κυβερνήση να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Θα περιοριστώ σε αυτά προς το παρόν. Έλπιζω να σας άνοιξε την όρεξη για συζήτηση, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ε, κύριε Πρόεδρε, είμαι στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινούμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Λόγος θα κύριο Λίζε. Από το ΕΛΚ παρακαλώ όλους τους επόμενους πολιτές να περιοριστούν σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φιγκέρες για την εισαγωγή σας και για όλες τις προσπάθειες που γίνονται εν ώψη της διάστασης του Παρισίου από πλευρά σας. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστική αλλά και φιλόδοξη στρατηγική. Δεν μπορούμε βέβαια να θεωρήσουμε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα στο Παρίσι και ότι θα τα επιτύχουμε όλα μια μέρα μετά τη διάσκεψη. Θα είναι ένα μόνιμο καθήκον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βασικό είναι να το καταλάβουμε αυτό όλοι. Ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά για μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιτύχουμε αυτό το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου. Και αυτός ο στόχος πρέπει να συμπεριληφθεί και στο κείμενο. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να σας ενθαρρύνω εν ώψη αυτής της διάσκεψης να ε, ασχοληθείτε με τις αεροπορικές μεταφορές. Ξέρουμε τι καθήκοντα δώσαμε εν ώψη της διάσκεψης, αλλά δεν ξέρω πόσο προχωράει. Και για τις αεροπορικές μεταφορές διαπιστώνουμε ότι αν ε, είμαστε πολύ τυχεροί τα κράτη που συμμετέχουν στον ICAO, ICAO θα καταφέρουν να μην υπάρξει αύξηση εκπομπών που να μην αντισταθμίζεται. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας ως Ένωση, η Κομισιόν πρότεινε η βιομηχανία, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία τσιμέντου και χάλιβα, να μειώσουν μέχρι το 2020 ε, τις εκπομπές τους. Ενώ βλέπουμε λοιπόν ότι και οι αεροπορικές μεταφορές και οι μεταφορές μέσω των εσωτερικών ε, υδατίνων οδών ε, αντιμετωπίζονται πολύ γενναιόδωρα. Πρέπει οπωσδήποτε και εδώ να μπει η λέξη μείωση. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για αντιστάθμιση και σταθεροποίηση. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας μόνο με σταθεροποίηση, χρειαζόμαστε μείωση. Το κλίμα χρειάζεται μείωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από τους, σοσιαλιστές, Γκροτέ. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι θέλουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, όλοι θέλουν να εγκρίνουν ψηφίσματα, να, να καθορίζουμε τη διεύθυνση, αλλά ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Το πνεύμα μεν πρόθυμο είδε σάρξα ασθενής όπως λέμε. Ελπίζω να μην ισχύσει στο Παρίσι. Ο Πέτερ Λίζε ασχολήθηκε με τις, εναέρες, με τις αεροπορικές μεταφορές αλλά και για τις θαλάσσιες μεταφορές θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρξουν ρυθμίσεις και αντιμετωπίσαμε μεγάλες αντιστάσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι εσύ θα μας βοηθήσετε για να υπάρξει πρόοδος. Να ασχοληθώ όμως με κάτι άλλο. 20 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας προσπαθούν να ξεφύγουν, να διαφύγουν από πολέμους, άλλες καταστροφές και από ό,τι μας λένε εμπειρογνώμονες όπως ο κύριος Μάιερς από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ο αριθμός των κλιματικών προσφύγων θα ανέβει τα επόμενα χρόνια στα 200 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Οπότε πόσο λαμβάνετε υπόψη σας αυτό στην προετοιμασία των διεθνών συμφωνιών. Το συζητάτε, Εάν δεν ε, αλλάξουμε την κατάσταση του κλίματος, θα οδηγήσει πολλούς στις φτωχότερες χώρες, ιδιαίτερα της Αφρικής, να εγκαταλείψουν τις χώρες τους. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή και όλος ο τομέας της εμπορίας ε, εκπομπών. Επίκειται η μεταρρύθμιση μετά την ε, διάσκεψη για το κλίμα. Είδαμε την πρόταση της Κομισιόν, καλή και ισορροπημένη τη βλέπω. Αλλά τι ρόλο θα παίξει η Ευρώπη γιατί ορισμένοι από μας λένε δεν κάνει αρκετά η Ευρώπη ενώ άλλοι θεωρούν ότι θίγουμε την ανταγωνιστικότητά μας και κινδυνεύει η βιομηχανία μας. Πώς εκτιμάτε εσείς που είστε απ' έξω τις προσπάθειες της Ευρώπης, πώς τη βλέπετε από μακριά. Ευχαριστώ για το ECR, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Κυρία Φιγέρας, χαίρομαι που ήρθατε, ευχαριστώ. Μια ερώτηση για τη διαδικασία στο Παρίσι. Ξέρουμε ότι προχωράμε αργά, ότι πρέπει να επιταχύνουμε, επιταχύνουμε μετά επιβραδύνουμε, έτσι φαίνεται τουλάχιστον για τους εξωτερικούς παρατηρητές, αλλά φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά στον στόχο χάρη στην ασκούμενη πίεση. Έχουμε πέντε ημέρες για διαπραγματεύσεις πριν από την έναρξη. Ε, λοιπόν, οι τεχνικές συζητήσεις, πώς τις βλέπετε, οι διαπραγματευτέ ε, ακολουθούν την πρώτη που έχει επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο, έτσι ώστε και τεχνικά όταν πάμε στο Παρίσι να είμαστε σχεδόν έτοιμοι, να είμαστε κοντά, ώστε να υπογράψουμε μια συμφωνία με συνοπτικέ αν γίνεται διαδικασίε. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Από του ελεύθερου Χρυσάντε. Πρόεδρε, Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Φιέρας που ήρθατε. Εγώ θα ψήφισα υπέρ όλων αυτών που είπατε για το Παρίσι. Κάντε μια δήλωση, η οποία ήταν εύστοχη, η οποία μας εμπνέει. Τώρα για τις εθνικές συνεισφορές. Είπατε ότι καλύπτουμε το 70% του πλανήτη όσον αφορά τις εκπομπές συνδοξιδίου του άνθρακα εάν η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη συνταχθούν από την ίδια μεριά, καλύπτουμε σίγουρα ένα μεγάλο μέρος αυτό του 70%. Η ερώτηση μου αφορά τις άλλες μεγάλες χώρες υπεύθυνες για εκπομπές που θα γίνουν και ακόμα μεγαλύτερη εκπομπή στη Βραζιλία και η Ινδονησία συγκεκριμένα. Οι κυβερνήσεις τους έχουν ενημερώσει την διάσκεψη ως ε, προς το κατά πόσον και πότε θα υποβάλουν τις συνεισφορές τους, τις εθνικές τους συνεισφορές. Εγώ προσωπικώς ανησυχώ, διότι δεν βλέπω και πολύ πρόοδο εκεί. Έχετε κάτι να μας ενημερώσετε. Και κύριε Πρόεδρε, το θέμα της χρηματοδότησης. Εκατό δισεκατομμύρια απαιτούνται μετά το 2020. Κάπου πρέπει να τα βρούμε. Πώς ε, συνδυάζεται αυτό με τις εξελίξεις στο Παρίσι. Πολύ μάλλον καθώς από πλευράς προϋπολισμού εδώ έχουμε να κάνουμε με μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις ε, για τις οποίες οι χώρες δεν έχουν κονδύλια να διαθέσουν. Ευχαριστώ. Γκουέ. Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω λίγο την κυρία Φιγκερές που ήρθε σήμερα για να συζητήσουμε. Έχω μεγάλη εκτίμηση για το θάρρος που έχετε δείξει, την ενεργητικότητά σας, για τις προσπάθειές σας να αντιμετωπίσετε αυτό το κουτί της Πανδώρας. Το είπαν και άλλοι βεβαίω. Το βέβαιο είναι ότι εκτό από το έθνη χρειάζεται και συνεισφορά άλλων. Υπάρχουν χάσματα τα οποία πρέπει να γεφυρωθούν. Και ναι, λοιπόν, χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη συμφωνία για να μην καταστραφεί ο κόσμο. Η Επιτροπή Γιούνκερ δήλωσε ακριβώ αυτό την περασμένη εβδομάδα. Η επόμενη έξοδος μεταναστών θα οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να υλοποιούμε το πακέτο του Μπαλί και τη Τόχα του 2012. Πρέπει οι πλούσιες χώρες συναφώς να βοηθήσουν τις φτωχότερες χώρες, να βοηθήσουν και αυτές. Εδώ λίγα πράγματα έχουν γίνει. Πρέπει λοιπόν να αναβιώσουμε, να αναστήσουμε αυτήν την προσέγγιση. Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της προσπαθειάς μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Λέει ένας κανόνας ότι αυτοί που ηγούνται πρέπει να μαθαίνουν από τα λάθη τους και να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις των σφαλμάτων τους. Λοιπόν, εμείς ως δυτικός κόσμος αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και με την ευκαιρία να πω κάτι για την TTIP, τη συμφωνία TTIP, όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, το κομμάτι του περιβάλλοντος δεν έχει καταλήξει η συμφωνία όμω με τον Καναδά, η συμφωνία με τον Καναδά ολοκληρώθηκε και η σχετική έκθεση για το περιβάλλον είναι σαφέστατη. Θα έχουμε πιο εντατική παραγωγή, ε, κρέτος, περισσότερες μεταφορές, μεγαλύτερες επιπτώσεις στο κλίμα. Δεν ξέρω, αυτό ε, θα καταρριφθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Φιγέρες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για άλλη μια φορά, εκτιμούμε πάρα πολύ τι ήρθατε εδώ, είστε τόσο απασχολημένοι. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, μια-δυο ερωτήσεις στα επιμέρους βήματα αυτά που είναι πιο καθόδια για την Ευρώπη και πες να μας πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις τι οποίε θα πρέπει κάπω να τοποθετεί η Ευρώπη πρώτα πρώτα για την, ε, ε, την διαδικασία αυτή για τα βασικά θέματα διαπραγματεύσεις. Τι γίνεται με αυτές τις τρέχουσες ε, υποσχέσεις για τους δύο βαθμούς των INDC παρά το ότι όλες οι μόνο για τους δύο βαθμούς ότι θα πρέπει να κατέβουμε. Και ξέρουμε ότι αυτή δεν θα είναι εύκολη διαδικασία, να δούμε πώς όλα αυτά τα μεταφράσουμε στη γλώσσα της Συμφωνίας των Παρισίων, γιατί πάντοτε η Ευρώπη δυσκολεύεται όσον αφορά το μήκος της ε, περίοδου διάσμευσης γιατί μόλις καταλήγουμε σε κάποιο ποσοστό τότε αυτό που θέλουμε είναι να ισχύσει αυτό για μια δεκαετία, κάτι το οποίο δεν φτάνει. Αλλά από παιδιά πρωτοκόλλο του Παρισιού, μάλλον χρειάζεται μια περίοδος δε μέσα στις πενταετής, οπότε ε, να πάει η Ευρώπη για έναν στόχο του 2025 και να μην έχουμε βάλει το 2030. Άρα εσείς πώς βλέπετε αυτή τη θέση της Ευρώπης που έχει ορίζοντα το 2030. Γιατί ξέρουμε τι θέσεις έχει τώρα η Ευρώπη. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει κάποιος πιο φιλόδοξο στόχο πριν το 2030, αλλά κανεί δεν το λέει αυτό στην Ευρώπη, γιατί θα ανοίξει τότε το κουτί της Πανδώρα. Οπότε, αν να έχουμε το 2030 ε, και να ξεχάσουμε φιλοδοξίε της Ευρώπης για το 25. Άρα για αυτή την ε, περίοδο δέσμευσης της πενταετίας πώς το βλέπετε πώς θα μπορούσε να ξυπνήσει νωρίτερα η Ευρώπη αφού βλέπει το το ώρα πλευράς χρηματοδότησης ανέκαθεν λένε οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχουν χρήματα και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε συμμετοχή και του δημοσίου του ιδιωτικού τομέα, αλλά πολλέ αντισώμενες χώρε στο Παρίσι προσβλέπουν στην Ευρώπη για χρήμα το δημόσιο τομέα και θέλουν κάτι σταθερό, δεν θέλουν να κλείσονται κάθε χρόνο όπως ισχύει τώρα, επομένως να μην κρύβεται πια η Ευρώπη και να λέει κάθε χρόνο, ε, να υπάρχουν 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο κλπ. Όμως ε, θα πρέπει τη οι Υπουργοί Οικονομικών μας να ασχοληθούν σοβαρότερα με το θέμα αυτό, γιατί τώρα θυμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η FTD. πια Νικόλα Πεντιτσίνη. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε και κυρία ε, Φιγέρης που ήρθατε να μας δείτε σήμερα. Αυτό ακριβώ που αναφέρετε προηγουμένω, ξέρουμε ότι όλε οι αντισώμενε χώρε θέλουν μια αναθεώρηση ε, επί τη βάση του IMDC για το διοξείδιο άνθρακος, αλλά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πλούσιες χώρες που είναι η βασική πηγή των εκπομπών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή κάθε δεκαετία, λέμε, οπότε είναι τέτοιου είδους δέσμευση τώρα που δεν είναι αρκετή όσον αφορά αυτό το 2% που βάλουμε το 2050 Οπότε το COP21 θα αναβαγίσει εάν δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση παληθεύσιμη, ε, δεσμευτική, προβλέψιμη κλπ. Τώρα να σταθώ συγκεκριμένα σε αυτή την ε, πολιτική πάυση χρήση του άνθρωπος γιατί καταλήγουμε σε ένα διοξείδιο του άνθρωπος το οποίο εκπέμπεται στον, στην ατμόσφαιρα από όλη τη χρήση ε, των, των καυσίμων και φτάνουμε σε, φόβο σε δύο, σχεδόν τρία εκατομμύρια τόνους. Οπότε αυτό το 2% αντιστοιχεί σε, πολύ λιγότερες εκπομπές. είμαστε επομένως στο 50 φορές ε, περισσότερες εκπομπές από ό,τι φροντίζουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα κατά τη γνώμη μας δεν είμαστε σωστό δρόμο. Θα πρέπει να σταματήσουμε τα ορυκτά καύσιμα και να έχουμε κάποιες λύσεις να μην είναι ευαλωματικές οπότε θα πρέπει να σταματήσουμε να αναβάλουμε συνέχεια και να το κλειοδοτούμε το πρόβλημα στις μέλουσες γενναίες και έτσι να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια μέτρα για να σταματήσει οι εκπομπέ του άνθρακα με δεσμευτικό τρόπο. ΕΝΕΦ. Ντορνανό. Ε, σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γραμματέα που ήρθε να μας δει. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η προβληματική και κυρίως γιατί και εμείς εδώ έχουμε εγκρίνει ένα σωρό νομοθετικά κείμενα τα οποία έχουν επιπτώσεις άμεσα σε εκατομμύρια και εκατοντάδε εκατομμύριων. Είναι στρατηγική σημασία στο θέμα. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλές διαφορετικές χώρες. Αυτό θέλω να τονίσω. Στη ΣΥΠΑ μπορούν να συντονιστούν για μια πολιτική κατά του κλίματος. Αλλά έχουμε πολλές χώρες που διαφέρουν πάρα πολύ όσον αφορά την οικονομία τους. Άρα πώς θα αγγίξουμε σε αυτές τις χώρες ε, αφού η οικολογία φρενάρει την πρόοδό τους. Επομένως, ε, Πρόεδρε, πώς να ελπίσουμε να υπάρχει μια πραγματικά ε, παγκόσμια συμφωνία όταν δεν θέλουν να δεσμευτούν οι βασικοί οι οποίοι μολύνουν, έχουμε όλες αυτές τις αρνητικές στάσεις εδώ στην Ευρώπη από διάφορα κράτη. Οπότε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτές τις εκπομπές ε, που φέρουν το πνεύμα του θερμοκηπίου τη ρώτησα και τίποτη για το 9,2% της ε, μείωσης μεταξύ 8 και 12 θα έχουμε 2,4% μείωση που προέρχεται επειδή το ΑΕΠ της Ένωσης έχει μειωθεί. Οπότε ε, θέλουμε μια πράσινη ανάπτυξη και ο εθνικός πλούτος να μην βλάπτει το περιβάλλον. Αλλά βέβαια δεν θέλουμε η οικονομική κρίση να κάνει καλό στο περιβάλλον αλλά να κάνει κακό στο, στον κόσμο και στην οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει ο και τώρα κύριε Φιγγέρες, έχετε το λόγο για τον πρώτο γύρο απαντήσεων. Πολύ αυτοκές οι ερωτήσεις. Να τις ομαδοποιήσω λίγο. Ξεκινώ την τελευταία ερώτηση. Γιατί είμαι βέβαια ότι ξέρετε πως ε, όλες οι χώρες καλύπτονται και όχι ορισμένες. Και όλες οι χώρες συνεχίζουν να έχουν δεσμευτεί σε αυτήν την συμφωνία ακριβώς με την διαδικασία που περιγράψατε. Να μειωθεί το GHG και να αυξηθεί η ανάπτυξη. Άρα αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Αυτό είναι στο επίκεντρο της Συμφωνίας των Παρισίων. Για να δούμε τώρα κάποιες ερωτήσεις για συγκεκριμένες χώρες και μετά να δούμε τις γενικότερες ερωτήσεις. Η ένδυση από Βραζιλία, η Ινδονησία, έχουμε τη δέσμευση της 27ης 12 η Ινδία και η Ινδία, η Ινδία η 27 Σεπτεμβρίου τελευταία. Η Ινδονησία θα προσχωρήσει τώρα, σύντομα, χωρίς να έχουν πει συγκεκριμένη ημερομηνία. Όμως έχω την αίσθηση ότι οι χώρες του G20 θα καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε να τηρηθεί η προθεσμία του Οκτωβρίου και έτσι να συμπεριληφθούν στην συνθετική έκθεση της πρώτης ενδεκάτου. Η Ινδία, όπως ρωτήσατε, πολύ σημαντική χώρα. Δεν ρωτήσατε για την Κίνα, αλλά και η Κίνα θα υποβάλει το εθνικό πρόγραμμα NDC. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση η Κίνα λόγω, η Ινδία λόγω των διαφορών της με την Κίνα. Και αυτό να το προσέξουμε. Και ξέρουμε τι πρεσβεύει ο Πρωθυπουργό της Ινδίας σε σχέση με την συνάντηση κορυφής. Οπότε θέλει να υπάρχει μια αγορά βασιζόμενη στη ζήτηση για τις χώρες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν αυτό που θα απασχολήσει την ε, συνάντηση κορυφής για την ηλιακή ενέργεια. Να καλυφθούν 15 μοίρες πάνω τον Ισημενό, 15 νοτίως, οπότε τέλος πάντων η προσέγγιση του είναι τεχνολογική πολύ διαφορετική από άλλες χώρες που βασίζουν στην πολιτική την προσέγγιση τους. Άρα πρόοδος της τεχνολογίας. Αυτή είναι η βάση της συνδικής πολιτικής. Βέβαια υπάρχουν και τα θέματα ε, πνευματικής ιδιοκτησία, τα οποία απασχολούν τους σύνδους, αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον η άποψή τους και να δούμε τι θα πούν οι άλλες χώρες. Δεν αναφερθεί στη συμφωνία με τον Καναδά. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό ας απασχολήσει εσά. Ε, όλο και κάτι θα μείνει για σας. Να, αυτό περισσεύει, ασχολείται εσείς. Η ΚΑΟ και ΑΕΜΟ. ναι, για τις καταθράσα και εναέριες μεταφορές, ξέρετε πώς είναι δομένη η συμφωνία, για εθνικές εκπομπές, γι' αυτό δεν καλύπτονται οι διεθνείς, ε, φυσικά και συνεργαστήκαμε και με τους δύο αυτούς οργανισμούς και βοήθη βοηθήσαμε στο έργο τους και τώρα εξαρτάζεται το πώς μπορεί να έχουμε κάποιο είδους παρεκκλήσεις αντί για μείωση για τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις τέλος πάντων από ό,τι ξέρουμε δεν πάνε για βραχυπρόθεσμη μείωση τέλος πάντων όχι πριν το Παρίσι οπότε να δούμε τι θα λέει η συμφωνία για να ενθαρρύνουμε περισσότερους οργανισμούς αυτούς να κάνουν μειώσεις. Βέβαια, είναι και το θέμα της τεχνολογικής προσέγγισης, να έχουμε δυο καύσιμα για την ε, αεροπλοεία, αλλά και για τις καταθάλασσες μεταφορές. Θέλουμε να υπάρχει λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ε, σε αυτή τη φάση το σημαντικό. Αλλά στην επόμενη φάση θα έχουμε τις μειώσεις. Οπότε Εκεί μετράει αυτό το οποίο αναφέρεται τώρα. Τι θα κάνουμε με αυτό το οποίο ε, ονομάζω εξαναγκαστική, αναγκαστική μετανάστευση. Οδυνήρη κατάσταση, δύσκολο πρόβλημα, όπως διαπιστώσαμε. Έχουμε όλες αυτές τις ε, οδυνηρές φωτογραφίες στον τύπο. Έχουμε όλα αυτά τα σενάρια και κάθομαι και αυτό τα πολλαπλασιάζω 10, 100, 1000, εκατομμύριο φορές. Να, τι σενάριο θα πρέπει λέω να αποφύγουμε. Και υπάρχει μια ομάδα χωρών που στο σχέδιο κειμένου εκεί που λέει για ζημία αποζημίωση τέλος πάντων λέει για ποιου είδους θεσμική ρύθμιση μπορεί να γίνει για να ανασχέσουμε αυτήν όλη τη μετανάστευση να έχουμε κάποιο συντονισμό με φοβίζουν όλα αυτά γιατί εγώ με κάθε τίμημα θα ήθελα να αποφύγω κάτι έτσι. Όμως τώρα υπάρχει στο σχέδιο κειμένο. Αυτό πρέπει να δούμε. Και θα έπρεπε να δούμε πολύ πιο εντατικά τόσο ώστε να φρενάρουμε όλα αυτά για να μην φτάσουμε σε, σε επίπεδα προβλήματος που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Κάποιοι τα σκέφτονται έτσι. Για τα INDC σε σχέση με την περίοδο αναθεώρησης, πενταετία, δεκαετία, κατέβασαν τέτοια προγράμματα, προτάσεις για 20, 25, 30, κάποιες χώρες, άγνωστο τι θα κρυθεί τελικά, αλλά τι να σας πω, πρέπει να κοιτάξω τη μαγική σφαίρα για να προβλέψω τι θα γίνει για την περίοδο που κάθε χώρα έχει καθορίζει. Επομένως, ε, υπάρχει κάποιο αυτοπιθαρχία, αλλά υπάρχει μια ένα, μια συμφωνία όλων μαζί, δηλαδή ο καθένας κατεβάζει πρώτε θέλει, αλλά, αλλά η αναφιόρεση θα πρέπει να είναι αντικείμενο συμφωνία από όλου. Λοιπόν, αν κάποιο κατεβάσει δεκαετέ INDC, κάποιο, ε, για πενταετή περίοδο έχει δεσμευτεί να κάνει αναφιόρεση, Οπότε νομίζω ότι εκεί πέρα πάμε να καταλήξουμε σε αντίθεση με την δεκαετία. Τότε να γίνει η αναθεώρηση. Και η κουβέντα τώρα είναι ότι ακόμα και εκείνες οι χώρες που θα κατέβαζαν μια πρόταση για δεκαετία να έχουν την ευκαιρία να συμφωνήσουν ε, σε μια τέτοια περίοδο αναθεώρησης και όχι σε δεκαετή. Αλλά τέλος πάντων πίσω από αυτά τι κρύβεται. Το πνεύμα της συμφωνίας που είναι το πώς θα υπάρξει ευελιξία, πώς θα υπάρχει κάτι που θα διευκολύνει και δεν θα είναι τιμωρητικό. Δεν ξέρω επομένως κατά πόσον θα υπάρχει υποχρεωτική ρύθμιση. Να δούμε πού θα καταλήξουμε και πώς θα έχει το τελικό κείμενο. Όσον αφορά τα διαφορετικά επίπεδα εργασίας, αναφερθήκατε στο τεχνικό επίπεδο και το πολιτικό επίπεδο. Σημειώνω ότι είναι πρώτη φορά από το 2009 που η Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή είναι σε τρία επίπεδα. Όχι μόνο δύο. Τεχνικό επίπεδο με τους διαπραγματευτές, σε απευθείας πολιτικό επίπεδο με τους υπουργούς, αλλά επίσης και σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Και αυτό το έχει αναλάβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας και η Καγκελάριος Μέρκελ, ο πρόεδρος Ολάντ και ο πρόεδρος Ουμάλε του Περού. Αυτή η τετράδα ηγετών έχουν αναλάβει να απευθυνθούν σε όλους τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης αυτής της συμφωνίας. Δεν είναι κάτι για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό ανοίγει δρόμο για αρκετές δεκαετίες, αν όχι ετία. Γι' αυτό, επειδή θέλουμε πραγματικά να αλλάξει μακροπρόθεσμα την κατάσταση πραγμάτων, οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων, συμμετέχουν και τώρα θα είναι στο, στη Νέα Υόρκη τον ε, Σεπτέμβριο και 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου θα είναι στο Παρίσι. Για πρώτη φορά θα κληθούν από την πρώτη μέρα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όχι μόνο στο τέλος, ακριβώς για να υπάρξει αυτή η καθοδήγηση από το ανώτατο επίπεδο. Επειδή έχουμε λοιπόν αυτό το τριπλό επίπεδο, έχουμε και διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ των τριών αυτών επιπέδων. Επιχειρούμε όσο γίνεται δηλαδή να αποκομίσουμε ωφέλη από την αυξανόμενη συνένεση σε αυτά τα τρία επίπεδα στα επακόλουθα σχέδια κειμένου όπως προχωράμε. Σχέδια για από μείωση της χρήσης άνθρακα. Καλούμε τις χώρες να υποβάλουν σχέδια μείωσης χρήσης άνθρακα μετά την έγκριση της Συμφωνίας Άνθρακα. Αυτό δεν θα αποκλίνει τόσο πολύ από τα NDC, ε είναι απλώς θέμα πώς θα εφαρμόσει ο καθένας την εθνική του συμβολή. Είναι λοιπόν τμήμα των τεχνικών λεπτομεριών του πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία του Παρισιού σε εθνικό επίπεδο. Για το σχόλιο για τον αναπτυσσόμενο κόσμο να μάθει από τα δικά μας λάθη, ναι, αλλά ο αναπτυσσόμενος κόσμος βλέπει και την ευημερία που επιτέχει, ε, πέτυχε ο εκβιομηχανισμένος κόσμος μέσω της χρήσης φορικτών καυσίμων. Άρα δεν μαθαίνουν μόνο από τα λάθη μας, βλέπουν και τις επιτυχίες μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί κάθε αναπτυσσόμενη χώρα έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να χορηγήσει σε κάθε πολίτη στους, ε, την ευημερία που έχουμε, εντάξει δεν έχουμε όλη την ίδια, αλλά που γενικά έχουμε εμείς εδώ, στον αναπτυγμένο κόσμο. Και φυσικά έχουν δικαίωμα οι πολίτες και φυσικά έχουν υποχρέωση οι ηγεσίε να το πετύχουν, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη η πρόκληση. Οπότε περνάω ακριβώς στη χρηματοδότηση όλων αυτών. Κάποιος είπε κρυβόμαστε πίσω από μια έκθεση. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η έκθεση του ΟΣΑ θα βοηθήσει πολύ. Θα σημειώσει το επίπεδο στο οποίο είμαστε τώρα. Θα λάβει τα στοιχεία από τη μόνιμη Επιτροπή Χρηματοδότησης που μας λέει ποιες είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές ε, χρηματοδοτικές ροές. Η έκθεση ΟΣΑ θα μας δώσει πάνω κάτω τα ίδια για τις χρηματοδοτικές ροές 13-14 του ΟΣΑ για το 11-12. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση όσον αφορά τις χρηματικές ροές και από δημόσιες και από ιδιωτικέ πηγές. Μετά το καθόδε θέμα είναι και μετά τι γίνεται. Διότι να μην ξεχάσουμε τη δέσμευση όλων μας. 100 δις μέχρι το 2020 και δεν τα έχουμε. Τα τελευταία στοιχεία που είδαμε είναι πιο κοντά στα 40-50 δις αν τα συνυπολογίσεις όλα, δημόσια και ιδιωτικά. Άρα υπάρχουν ε, εύλογες προσδοκίες. Θέλουμε το Παρίσι να δείξει το δρόμο για το πώς από αυτά που έχουμε τώρα θα περάσουμε στα 100 το 2020. Τι είναι λογικό να περιμένουμε για το 16 δηλαδή, το 17, το 18. Τι είναι εύλογο να περιμένουμε. Και δεν είναι νομίζω παράλογες αυτές οι απαιτήσει. Γιατί αυτές οι ροές ήδη διαπιστώνονται. Έχουμε ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες, είναι όλο και πιο ενδιαφέρουσες επενδύσεις και βλέπουμε να γίνονται επενδύσεις, να αραίουν κεφάλαια προς όλα αυτά. Δεν είναι λοιπόν παράλογο να περιμένουμε να υπάρχει διαφάνεια, για τα ορόσημα που θέλουμε να επιτύχουμε στην πορεία προς τα 100 δις μέχρι το 20. Πώς θα τα βάλουμε τώρα όλα αυτά στο κείμενο. Ναι, δεν είναι εύκολο, το παλεύουμε. Γιατί η πληροφόρηση για τις επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις ε, είναι από πολλές πηγές. Πώς θα φτιάξουμε δηλαδή μία κεντρική πηγή για να έχουμε αυτά τα στοιχεία ούτω ώστε και στη συμφωνία και στα πορίσματα να υπάρχει δυνατότητα, να υπάρχει ένας χώρος όπου να μπορούν να συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες για τη χρηματοδότηση. Δεν έχω τώρα συγκεκριμένη απάντηση, αλλά είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντική προτεραιότητα να δούμε πώς να υπάρξει μια πολιτικά αποδεχθή, αποδεκτή αλλά και αποτελεσματική πηγή πληροφόρηση για τη χρηματοδότηση. Και α, ξέχασα την καλύτερη απάντηση που θέλω να σας δώσω. Πώς αντιμετωπίζεται από τα έξω η Ένωση. Η Ένωση αντιμετωπίζεται ως ε, αναμφισβήτητα η πιο φιλόδοξη, η πιο μεθοδική και η πιο υπεύθυνη δύναμη. Πολύ θετικά. Θέλω να το τονίσω αυτό. Η υψηλότατη εκτίμηση υψηλότατη εκτίμηση χέρι μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Εκτιμούν ιδιαίτερα το ρόλο που παίζει η Ένωση για να τραβήξει μπροστά την κατάσταση, ενώ ορισμένοι άλλοι φρενάρουν. Πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ λοιπόν των δύο τάσεων και η προωθητική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται πολύ από τις αντισώμενες χώρες. Πολλές αντισώμενες βέβαια θέλουν να κάνει περισσότερα, αυτό είναι κατανοητό, αλλά παίζει πραγματικά ρόλο ως πρότυπο. Ακριβώς επειδή καταφέρατε να αποσυνδέσετε το ΑΕΠ από τα επίπεδα αερίων θερμοκηπίου. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε και στις αντισώμενε χώρες ότι αυτά τα δύο μπορούν να αποσυνδεθούν. Θα βοηθούσε πολύ να το καταλάβουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Παρακαλώ τους συναδέλφους να τηρούν ε, χρόνο ενός λεπτού, γιατί έχουμε 18 συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Να ξεκινήσω με τον Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Φιέρης. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, Μίλησατε για το ευρωπαϊκό παράδειγμα και ο Σάνθος Γκρότε αναφέρεται το ETS σύστημα, το σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών στην Ευρώπη. Το σώσαμε το σύστημα αυτό χάρη στο αποθεματικό σταθεροποίησης της αγοράς. Θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες το σύστημα αυτό και στο Παρίσι θα παίξει κάποιο ρόλο εάν νομίζω ότι μπορεί να παίξει ρόλο. Για την οικονομική βοήθεια τώρα, αναφερθήκατε στην Ινδία, στην μεταφορά τεχνολογία, ωραία πράγματα όλα αυτά. Βεβαίω. Όμω υπάρχει και η μεταφορά τεχνολογία, η οποία και αυτή πρέπει να γίνει. Για τον ΙΚΑΟ τώρα στι αερομεταφορέ, δεν περιμένουμε συμφωνία σύντομα. Πώ βλέπετε την αντιστάθμιση των εκπομπών σε διεθνεί πτήσει. Εγώ το κάνω αυτό πετώντα το Στρασβούργο κάθε φορά μια φορά το μήνα, πληρώνω 10 ευρώ. Δεν είναι πολύ. Θα μπορούσαμε να ανισταθμίσουμε ακόμα και σε επίπεδο τεράστιων μεγάλων πολυεθνικών εταιριών ή είναι ουτοπικό αυτό να το περιμένουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πάνια. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε, ευχαριστώ για τι απαντήσει σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Εγώ είμαι εισηγητή εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το κείμενο πρωτοβουλία για την COP21 με τίτλο προ μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα. Στο Παρίσι φυσικά. Να σα πω εντάχει σε λίγο τρόπο ένα λεπτό γιατί και πώς ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουμε σε αυτό το μοντέλο, σε αυτήν την φιλόδοξη προσπάθεια ακριβώς όπως το είπατε. Γιατί από της εικόνε που θέλουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή συζητούμε τροπολογίε, συμβαστικέ τροπολογίε. Ε, πιστεύουμε ότι πρέπει όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει κατά τουλάχιστον 40% στο 2030 τι εκπομπές της. Να μειώσουμε 30% την κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση μας, την ενεργειακή μας απόδοση, να την βελτιώσουμε και αυτή κατά 40%. Αυτό μέχρι να ακολουθήσει και ο πλανήτης ε, το 2050. Χαίρομαι πολύ που η περίοδος δέσμευσης είναι πενταετής, κάτι το οποίο θα μας επιτρέπει να αξιολογούμε σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα και θα να τροποποιούμε τις δράσεις μας για να αντιμετωπίσουμε τη μεταβολή του κλίματος. Και κάτι άλλο, τα οικονομικά. Το οικονομικό κομμάτι που είναι ακρογωνίως λίθος τη συμφωνία που θα αρχίσουμε να συζητούμε στο Παρίσι τέλη Νοεμβρίου, αρχέ Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να μα πείτε λίγο περισσότερα όσον αφορά την καινοτομία που, που απαιτείται για να εξασφαλίσουμε τα περίφημα αυτά 100 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Πρόεδρος Τάνκαν. Κύριε Φιγέρες, εδώ είμαι στη μέση. Ευχαριστώ που ήρθατε στην Αυστραλία έμαθε τι έγινε. Άλλαξε η κυβέρνηση και μάλιστα ερειπεί ο Κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγή πολιτικής που μας υπενθυμίζει όχι μόνο τις δυνατές θετικές εξελίξεις αλλά και τις ενδεχομένες αρνητικές. Γιατί δεν αλλάζουν μόνο οι κυβερνήσεις. Δεύτερον, η κατάσταση στην Κίνα. Υποτίθεται ότι οι εκπομπέ του θα κορυφωθούν το 2030. Φορά απογοητευτικό, δηλαδή πού πάμε. Μήπως θα πρέπει να έχουμε ένα πιο φιλόδοξο στόχο για την Κίνα. Επόμενος βελητής. Πρόεδρε, συζητούμε την μεταβολή του κλίματος. Σε τέτοιες συζητήσεις δύο προσεγγίσεις προκύπτουν. Η μία συνιστάται στην προσπάθεια να πείσουμε τα κράτη, τα κράτη να κάνουν κάτι και από την άλλη μεριά προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά σε εισόδημα κατά κεφαλήν γιατί μια χώρα έχει 5 εκατομμύρια πληθυσμό η άλλη μπορεί να έχει σε λίγο 5 δις ευθύνη για το περιβάλλον είναι βεβαίως πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ισοποδοτικές λύσεις. Και εκτός από τα κοινά μας συνέθλια έχουμε, ελπίζω και αυτό το κοινό κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Φιγκέρες που ήρθατε θαυμάζω την αισιοδοξία σας, αν και δεν τη συμμερίζομαι. Θεωρώ ότι η μείωση των εκπομπών και ο περιορισμός ε, της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι δύο βαθμούς από τη μία και αυτό το μάντρα για συνέχιση της ανάπτυξης από την άλλη ως ε, τετραγωνισμό του κύκλου. Και όπως ε, συχνά έχω πει στο σώμα εδώ, αυτή τη στιγμή έχουμε παραγωγή κρέατος 300, 300, 300 εκατομμύρια τόνους και μας λένε ότι σύντομα θα αυξηθεί. Τι σκοπεύει να κάνει ο, Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τις εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή κρέατος. Θα ληφθούν υπόψη αυτές οι εκπομπές ή το θέμα του κρέατος άλλη μια φορά θα το αφήσουμε κατά μέρο γιατί είναι νόστιμο το κρέας. Και θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος δεν μαθαίνει ποτέ τίποτα. Γιάβορ. Ε, Γιάβορ. Τρεις γρήγορες ρωτησούλες, Πρόεδρε. Συμφωνούμε ότι τα INDC πόρο απέχουν από το να πετύχουν το στόχο μας. Τι να κάνουμε, πώς να βάλουμε τον πύχη πιο ψηλά στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού. Μας είπατε τι γίνεται με τα σπάνια τρόφιμα, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει και τόσο πολύ. Πώ θα φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι θα κάνει ο Ιεούτος ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε μέσω της Συμφωνίας των Παρισίων ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιθαγενών και άλλων πληθυσμών. Δεν μιλάμε τώρα εν κενό για το κλίμα. Έχουμε και διαπραγματεύσει τον ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς θα εξασφαλίσουμε το να συνάδουν οι στόχοι της μείωσης των εκπομπών με τα υπόλοιπα. Πώς η συμφωνία το κλίμα μπορεί να μας βοηθήσει στους υπόλοιπους στόχους, πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε έναν βιώσιμο κόσμο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ο κύριος Έδει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ, εδώ είμαι. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι που το είπε ο συνάδελφος πριν γιατί θέλουμε να τραγουδήσουμε τον κύκλο δηλαδή να εξυπηρετήσουμε και την οικονομία και το περιβάλλον οπότε να δούμε μήπως μπορούμε να προεκτείνουμε το σύστημα εμπορίας των εκπομπών σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη γνώμη μας όμως το σύστημα αυτό ETS απεδείχθη αναποτελεσματικό στην Ευρώπη. Μια από μια δεκαετία, τέσσερι φορέ αναθεωρήσαμε τι διατάξει αυτέ και δεν απέδωσαν για τι εκπομπέ. Αντίθετα, έπληξαν την παραγωγή τη βιομηχανία και επίση έδωσαν έδαφο σε χειραγωγήσει, σε απάτε, κερδοσκοπίε. Είδατε στο Μιλάνο τι υποθέσει ε, δικάζει δικαιοσύνη. Οπότε Κάτι γνώμη σας. Τι να κάνουμε, να πρέπει αυτό το σύστημα να το υιοθετήσουμε, να το παρεκτείνουμε σε διεθνές επίπεδο ή να βρούμε το θάρρος να υιοθετήσουμε νέα πρότυπα ή νέους φόρους των ε, ρηπαντών με διοξίδιο του ε, άνθρακα. Η κυρία Ντάλη τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Φιγκερές που ήρθατε να μας δείτε. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή των απόψεων και ήταν θετικό αυτό που ακούσαμε. Ότι είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτη σε αυτό το περίπτωση ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε συγκεκριμένου τομεί προβληματιζόμαστε. Εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε τι γίνεται με τον Λιγνίτη. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Λιγνίτη τώρα. Έχουμε 10% εκπομπές και πάνω προέρχονται από εκεί. Επίσης, βλέπετε, έχουν λιγνητορυχία και, και διάφορες σχετικές καταστάσεις και μιλάμε για ε, διάρκεια ζωής πάνω από 40 έτη. Επιδοτούνται κάποιες εταιρείες που παίρνουν άνθρακα από το εξωτερικό Εκεί μιλάμε για 40% των εκπομπών παγκοσμίω που έρχονται από τον άνθρακα. Οπότε τελικά δεν είναι θέμα της Υπήρου, δεν είναι θέμα μιας χώρας, είναι παγκόσμιο. Άρα οι χώρες δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να εξάγουν την ε, μόλυνση στο εξωτερικό. Εσείς τι λέτε, τι διατυπώσατε, τι, τι διαπιστώσατε μέχρι τώρα. Δεν πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Thank you very much. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Λαβία. Η κυρία Βυσνιεύσκα έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σίγουρα η Επιτροπή αυτή θα συμφωνήσει ότι πρέπει να πάμε σε μείωση των υπομπών μέχρι το 2030 κατά 40%. Και έτσι με το δεξί θα ξεκινήσουμε τις θερμοτέρες στο Παρίσι τώρα. Ποιες θα είναι για όλη την Ιφίλιο ε, οι συνέπειες, μια που έχουν αναλυφθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Είπαμε ότι θα πρέπει σε σημαντικό βαθμό να μην ζεγμομπέσει η Ένωση. Αλλά τι γίνεται σε Κίνα, Ινδία και είπα. Εμείς θα κάνουμε τις μειώσεις. Αλλά θα πρέπει να έχει αυτό επιπτώσεις στην παγκόσμια σκηνή, άρα δηλαδή και οι άλλοι να κάνουν αυτό που κάνουμε και εμείς. Μήπως θα πρέπει να έχουμε δεσμεύσεις συγκρίσιμες και αυτούς τους άλλους ρηπαντές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέντρελε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φιγκέρες για τις θαυμάσιες παρατηρήσεις σας και τις σαφέστατες απόψεις σας για τις διαπραγματεύσεις. Είμαι Σουηδός. Και η Ευρώπη παίζει ηγετικό ρόλο και εμείς ως Σουηδία παίζουμε ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. Εμείς εξετάζουμε την κατάσταση και το κόστος της αν δεν κάνουμε τίποτα. Τι συνέπειες θα έχει για δημόσια υγεία, τον προϋπολογισμό μας, ε, τη γη μας που θα πάει στράφη που αυτή τη στιγμή παράγει κτλ. Για να καταλάβουμε το διακύβευμα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ποιες θα είναι οι πλανητικές αλλά και περιφερειακές και εθνικές επιπτώσεις για να καταλάβουμε και τι επενδύσεις πρέπει να κάνουμε, τι ύψους επενδύσεις και, και τι είδους επενδύσεις. Όσοι δεν θέλουν να κάνουν σωστές επενδύσεις μιλάνε μόνο για το κόστος. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 η, η Σουηδία συγγνώμη, έκανε αυτή την αποσύνδεση μεταξύ εκπομπών άνθρακα και ανάπτυξης και έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ανάπτυξης από τα υψηλότερα στον κόσμο μειώνοντας εκπομπές. Παρ' όλα αυτά πολλά ακόμη πρέπει να κάνουμε αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει θα βοηθήσει νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες τεχνολογίες και θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να το δούμε από αυτή την οπτική γωνία. Νέε επενδύσει, ε, νέε θέσει εργασία. Μόνο έτσι θα επιτύχουν οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Τόρλα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να επιμείνω σε κάτι που δεν έχει τονιστεί αρκετά γιατί για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής μας. Είναι επίγον να κάνουμε 180 μοίρες στροφή στον τρόπο της οικονομίας μας, τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Πρέπει να μειώσουμε και με τον τρόπο λειτουργίας ε, των πόλεων και τις συγκοινωνίες ε, και εμένοντας στην, ε, στις ανανεώσιμες ενέργειες να επιτύχουμε ε, ένα νέο τρόπο οργάνωσης των δικτύων που να μειώσει και την ε, φτώχεια, την ενεργητική που φύγει το 10%. Και ο λόγος για την κλιματική αλλαγή είναι η καύση ορυκτών καυσίμων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί να αναπτύσσει το πλανήτη με ένα τέτοιο τρόπο. Ε, οφείλεται και στον τρόπο των δοσοληψιών αυτών των εκπομπών που επιτρέπει όποιο είναι πιο πλούσιο, να έχει το δικαίωμα να μολύνει περισσότερο Του πάντε θίγοντας και την υγεία των πολίτων ενώ οι ελίτ συνεχίζουν να πλουτίζουν. Η καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή σημαίνει θάρρο. σημαίνει πολιτική βούληση, σημαίνει εφαρμογή πολιτικών που να προωθούν υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη, υπεύθυνη για τον πλανήτη και του πολίτε. Όλα τα άλλα, εάν δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά τα δύο, μα βρίσκουν αντίθετους. Κατηγορηματικά αντίθετος. Ευχαριστώ. Η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Θαυμάσια παρουσίαση. Είχα ακούσει πόσο καλοί είστε. Τώρα όμως που σας άκουσα βλέπω ότι πραγματικά είστε όσο καλοί μου λέγανε. Και χρειάζεται να είστε καλοί γιατί χρειαζόμαστε ρεαλιστικά μηνύματα. Πολλοί πολιτική το αντιμετωπίζουν σαν να διαπραγματεύονται με τη φύση. Δηλαδή να μας δώσει αυτά η φύση για να τις δώσουμε εμείς αυτά. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα ήθελα οι ηγέτες μας να είναι τόσο σαφείς όσο το Πεντάγωνο και το ΝΑΤΟ. Που ξέροντας ότι οι συγκρούσεις ε, προκαλούν πρόσφυγες μας λένε τι πρέπει να κάνουμε για τις συγκρούσεις. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε όχι μόνο για τα θετικά που αναφέρατε για τα κράτη-μέλη και την Ευρώπη. Να εκτιμήσετε τι ρόλο παίζουν και τα αρνητικά μέτρα. Για παράδειγμα, η, η ε, Ναι, η αποθήκευση άνθρακα. Πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Γιώ Λάινεν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε Κριστίνα Φικέρες. Κάθε φορά που σας βλέπουμε σας ε, καλωσορίζουμε. Επανειλημμένα σας έχω δει και πάντα είστε πολύ αισιόδοξοι. Τώρα μας είπατε ότι περιμένω ότι η θα γίνει χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς ε, κλάματα και δράματα. Δεν το υποσχέθηκα, λέει η κυρία Α, εντάξει, να δω αν θα αγοράσουμε τη σαμπάνια και να μου πείτε αν θα μείνουμε στο ξενοδοχείο μόνο Παρασκευή ή πρέπει να το κλείσουμε και Κυριακή και Σάββατο. Ας ελπίσουμε λοιπόν. Αλλά εάν τελειώσετε νωρίς, ε, τη σαμπάνια την έχω ήδη πάρει, θα την πιούμε. Είπατε ότι η φιλοδοξία μας είναι το δεύτερο ήμιση του 21ου αιώνα να, η ανάπτυξή μας να είναι κλιματικά ουδέτερη. Πότε θα γίνει αυτό, το 2100? Ο στόχος μας είναι το 2050 να είναι κλιματικά ουδέτερη η ανάπτυξη. Τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν μείωση 60%. Ξέρω ότι οι Κινέζοι δεν συμφωνούν, αλλά υπάρχει κάποιο στόχο για το 2050 που θα μπορούσε να συμφωνηθεί στο κείμενο της ΚΟΠ. Ναι, βέβαια, η χρηματοδότηση θα είναι το τελευταίο και το μεγαλύτερο θέμα που θα πρέπει να επιληθεί κάποια στιγμή. Αυτά τα 100 δις μετά το 2020. Πολλοί το ρωτάνε. Θα είναι δύσκολο οι Υπουργοί Οικονομικών να δεσμευτούν για τις κυβερνήσεις τους μετά το 2020. Υπάρχει τίποτα για το πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα 100 δις μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων κατά την περίοδο 2020-2025 έως και 30 πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Σεπ Ντάνς. Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε κύριε Φιγέρες. Σας βλέπω αφοσιωμένοι στο στόχο σας όσο ήσταν στην Λίμα, φαραστική δουλειά κάνατε. Δείξετε ηγετικές ικανότητε που θα αποφέρουν καρπούς πιστεύω πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και που μα εξηγείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Όσον αφορά τη συμμόρφωση, καταλαβαίνω ότι συλλογικά μπαίνουμε σε ένα σύστημα προαιρετικό, όχι υποχρεωτικό, όσον αφορά του στόχου. Το κατανοώ αυτό σε διεθνέ επίπεδο. Έτσι, διαφορετικές χώρες θα κινηθούν με βάση τις διαφορετικές τους παραδόσεις, ο, συστήματα οργάνωσης κλπ. Τώρα όσον αφορά τις βασικές δεσμεύσεις έχουν γίνει βάσει της Κανκούν του 2010 όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όμως οι φυστάμενοι μηχανισμοί, η καθαρή ανάπτυξη, τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης της μεταβολής του κλίματος κλπ. Τα μέτρα μετριασμού δηλαδή. Αυτά επιτρέπουν στις ε, ΜΚΟ, για παράδειγμα, στην κοινωνία των πολιτών να πιέσουν ακόμη περισσότερο τις κυβερνήσεις τους. Πάμε στους επόμενους μελητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Εδώ, εδώ είμαι. Κυρία Φιγέρες, θα ήθελα περισσότερη ενημέρωση και διευκρινήση για δύο ζητηματάκια που στην αρχή θίξατε. Μας είπατε ότι θα είναι θέμα κλειδί η χρηματοδοτική υποστήριξη των επιστομένων χωρών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα όσον αφορά τη συνεργασία και ανάπτυξη για την εξωτερική πολιτική που καλύπτει τα θέματα αυτά, να δείξει αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ε, συνέπεια, αποτελεσματικότητα και λέω ε, συνέπεια γιατί, να, για παράδειγμα σε κάποια μέλη ε, οι επενδύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές αντί για αυτό το οποίο είπατε, αντί να προχωράει, ο πιστοχωρεί, μειώνεται. Οπότε για πετε μας, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι προσδοκάτε σε αυτό το μέτωπο τώρα όσον αφορά τις, ε, τα μη κυβερνητικά, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ε, τέτοιους φορείς. Είπατε ότι αναγνωρίζουμε το ρόλο τους, αλλά είπατε ότι είστε ικανοποιημένοι με τη θέση που έχουν σε αυτήν όλη την διαδρομή. Μα δεν θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να έχουν πιο σημαντικό ρόλο, πιο αποφασιστικά να παρέμβουν στις φάσεις όλες αυτές της διαδικασίας. Και έτσι μπορεί η συμμονή των Παρισίων να είναι πιο φιλόδοξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε. Τι γίνεται με, την, ε, με τα δάση και τη δασοπονία. Κανείς δεν μίλησε γι' αυτό. Τα δάση και στο βορρά και στο νότο διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα, όπως όλοι γνωρίζουμε. 10% των εκπομπών μας στην Ευρώπη δεσμεύονται από την δασοκάλυψη. Πρόσφατα συζητήσαμε μια στρατηγική για τα δάση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τη δασοκάλυψη, όμω δεν πρόκειται για δεσμευτική απόφαση και δεν έχουμε θέσει και ένα στόχο ποσοτικό, ένα ποσοστό. Καλό θα ήταν πάντω να αυξήσουμε τη δασοκάλυψη και όχι να καταναλώνουμε περισσότερα, περισσότερη ξυλία. Το ίδιο ισχύει και τον Νότο, το να μην εξαφανίζουμε τα δάση, να μην αποψηλώνουμε τα Βάση ήταν θετικό βήμα. η Νορβηγοί πλέον το, θα μπορούσαν πλέον το Περού για να μην κόβει τα δάση του. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αδελφοποιήσουμε έτσι, χώρες, ας πούμε Γερμανία με Βολιβία για να μην κόβει τα δέντρα η Βολιβία. Η... Το ίδιο με την Ουρουάη. Αυτό θα μπορούσε να προσθέσει κονδύλια στα κονδύλια που έχουν ήδη δεσμευθεί υπέρ της ε, Γνωστή υποθεση Να σώσουμε έτσι μερικά τάση. Η κυρία Κατενμπάχ. Επειδή αν υπομονώ να ακούσω τι απαντήσει σα, κυρία ε, δεν θα κάνω ερώτηση, έχετε τον λόγο αυτή, σε τι με αφορά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Φικέρες, πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της συνεδρίασης. Έχω 11 λεπτά μόνο. Δεν ξέρω αν πιέζετε τους παρά τους ομιλητές σας, αλλά ή τους πιέζετε με τόσες ερωτήσεις. Χαίρομαι για την πειθαρχία που έχει η συνεδρίασή σας. Λοιπόν, ξεκινώ με όλες τις ερωτήσεις που έχουν σχέση με τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση των προσπαθειών μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι ψάχνουμε για καινοφανή, καινοτόμα εργαλεία για να κρατήσουμε τις επενδύσεις πιο ασφαλείς. Γιατί τα κονδυλιά λείπουν, θα πώς θα τα επενδύσουμε με ασφάλεια στον εαυτό τομέα. Παρατηρούμε λοιπόν μια συνενωμένη δράση μεταξύ κυβερνήσεων, αναπτυξιακών τραπεζών, πώ το σκοπό αυτό. Επειδή με ρώτησαν, πείτε μου κάτι καινοτόμο, να σα πω, οι πολυμερεί αναπτυξιακέ τράπεζες διθέτουν περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία σώρευσαν κατά διάρκεια των δραστηριοτήτων τους από τότε που ιδρύθηκαν. Πώς θα αξιοποιήσουμε τα πόσα αυτά για να μπορέσουν να προβούν σε εκτεραμένο, πιο εκτεραμένο τουλάχιστον δανεισμό προς τις χώρες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις πολιτικές ε, μετριασμού και αντιμετώπιση της μεταβολής του κλίματος. Αυτό είναι μια ιδέα. Έχουμε τα πράσινα ομόλογα, για παράδειγμα, και έχουμε και άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Πάντω αυτή τη στιγμή όλοι αυτό κάνουν. Ψάχνουν να δούμε ποιο τρόπο θα χρηματοδοτήσουμε διάφορε τομεί όπω και τη δασοπονία μεταξύ άλλων. Εκεί η χρηματοδότηση είναι ένα από τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλοι συμφωνούμε προκειμένου και η συμφωνία πραγματικά τη Νορβηγία με το Περού είναι εξαιρετική. Η χρηματοδότηση πάντω αυτή θα εκταμιεύεται βάσει απόδοσης. Δεν τα δίνουμε τα λεφτά μπροστά, βάσει αποτελεσμάτων θα καταβάλλονται, θα πληρώνονται τα ποσά αυτά στο Περού συγκεκριμένα. Είναι ένα τεχνικό τομέα, ένα τεχνικό θέμα αρκετά σύνθετο, πάντως αποδεικνύει ότι υπάρχουν δυνατότητες πολύ καλής συνεργασίας βορρά-νότου. Είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένας από τους τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί πολύ καλή διεθνή συνεργασία. Έτσι κάπως φαντάζομαι την πρόοδο πω τα εμπρός και στον τομέα της χρηματοδότησης. Αυτό είναι σίγουρα μια πολύ καλή εξέλιξη. Καλή εξέλιξη δεν έχουμε για τη χρηματοδότηση μετά το 2020. Δηλαδή, το θέμα είναι, αν το έχετε ακούσει, τι θα κάνουμε μετά το 2020, γιατί ξέρουμε τι θα κάνουμε μέχρι το 2020, αλλά μετά το θέμα είναι εντελώ ανοιχτό, ούτε έχουμε ρίξει αρκετά το βάρος μας στο θέμα αυτό. Και εδώ θέλουμε την υποστήριξή σας, γιατί είπαμε μπορούμε να πάμε ικανοποιητικά μέχρι το 2020 και μετά να τα παρατήσουμε όλα. Δεν είναι αυτό το θέμα όμω. Οπότε και εδώ θα θέλαμε την υποστήριξή σας. Για τις εθνικέ συνεισφορέ. Η INDC ελπίζω ότι θα παραμείνουν αυτές που είναι αλλά και θα αυξηθούν. Γιατί είναι προ το εθνικό συμφέρον τη κάθε χώρα. Ξέρετε, δεν υποχρεώνουμε κανέναν να προτείνει κάτι. Ε, θέλουμε οι χώρε να προτείνουν κάτι το οποίο είναι προ το συμφέρον του. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο πιστικό από το ίδιο το εθνικό συμφέρον. Ελπίζω λοιπόν ότι οι αυτοί, αυτοί για τι εθνικέ συνεισφορέ θα υλοποιηθούν και θα υπερβαθούν για το καλό και τη κάθε χώρα Πρέπει να αντιληφθεί κάθε χώρα ότι είναι προ το δικό τη εθνικό συμφέρον να υλοποιήσει τον στόχο αυτόν, τον INDC. Γιατί η συλλογική προσπάθεια και η εθνική κατατείνουν προς, την... προς τον ίδιο στόχο. Συμφωνώ απολύτως με τον βουλευτή που είπε ότι είναι κατά των ισοπεδωτικών λύσεων. Όχι, χρειάζεται να δούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Χρειάζεται ευελιξία, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Σύμβαση των Παρισιών. Αυτό είναι και υπέρ και κατά. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να έχουμε αυστηρές απαιτήσει όσον αφορά τις, την υποβολή εκθέσεων, αλλά οι απαιτήσει, όπως είπα, είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. για την Κίνα. 2030 ναι, θα έχουμε για τον άνθρακα τις μέγιστες εκπομπές πριν αρχίσουν να μειώνονται. Αν ρωτήσει κανείς πότε θα αρχίσει να μειώνεται η καταναλωσία άνθρακα εκεί, θα σας έλεγαν ναι, δεν είναι και για αύριο. Πάντως ε, τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη άρχισε να μειώνεται επειδή έτσι είναι το εθνικό συμφέρον τη Κίνα, όχι επειδή το επέβαλε κάποιο. Α είναι καλά τα εθνικά συμφέροντα. Για το κρέα το κρέας δεν θα συμπεριληφθεί. Θέλω να καταλάβετε ότι η συμφωνία αυτή είναι μια γενική συμφωνία για τις επόμενες δεκαετίες. Ακόμα και η ενέργεια που είναι στην καρδιά του προβλήματος και η ενέργεια ε, μην νομίζετε ότι θα είναι αντικείμενο λεπτομερών ρυθμίσεων για τεχνολογίες κλπ. Αναφορά στο κράτο λοιπόν δεν θα γίνει. Λυπάμαι γιατί είμαι και χορτοφάγος, αλλά και στον τομέα αυτό παρακαλώ να, να συνταχθούμε από την ίδια πλευρά και να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας. Τρεις ερωτήσεις ακούστηκαν νομίζω. Α, από εσάς. Πώς σας έχασα. Πώς βρεθήκατε εδώ. στόχος είναι μεταβλητός. Οι στόχοι κινούνται συνεχώς, χτίζουμε πολιτικές συνενέσεις σιγά σιγά και προχωρούμε. Αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω εδώ και το οποίο είναι κρίσιμη σημασία είναι ότι πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον ποιος είναι ο τελικός στόχος για το δεύτερο μισό του αιώνα ουδέτεροι σε εκπομπέ, αλλά το πρώτο βήμα είναι η Σύμβαση των Παρισίων. Και μετά θα δούμε δικαιώματα του ανθρώπου. Λίγα πράγματα, γιατί το θέμα τη ισότητα των πολιτικών για την ισότητα των δύο φύλων, η μετάβαση για το εργατικό δυναμικό, τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών, όλα αυτά είναι κομμάτι της γενικότερη εικόνα, αν θέλετε. Είναι κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Δεν θα αναφερθούμε συγκεκριμένα σε τεχνικό επίπεδο σε όλα αυτά. Όμω η συμφωνία θα περιλαμβάνει αυτέ τι γενικέ προσεγγίσει, τι γενικέ αρχέ συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο συντονισμό με τι SDG θα έχουμε συνεργασία για το κλίμα αλλά και για την ενέργεια και την δασοπονία που σχετίζεται άμεσα με το κλίμα. Πιστεύω ότι λοιπόν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ενισχύοντας η μεν τους δε. Για τα εργοστάσια που καταλώνουν άνθρακα, να ξέρετε ότι όλο και περισσότερε εμπορικέ, τράπεζες και σίγουρα οι πολυμερείς αναπτύξεις τράπεζες, αλλά και οι χώρε ε, διμερώς, σταματούν τη χρηματοδότηση των ε, ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών που και είναι άνθρακα. Είναι μια τάση που προέκυψε τους τελευταίους 12 με 18 μήνες. Καλό αυτό, ε, γιατί καλό είναι να αφήσουμε τους ορεικτούς πόρους εκεί που βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Και νομίζω ότι ήταν άδικο αυτό που ακούστηκε, ότι δεν ακολουθούν οι άλλοι μεγάλοι εκπομπείς, οι μεγάλοι ρηπαντές. Ε, έχουμε 62 χώρες, παρακαλώ, που υπέβαλαν τις εθνικές τους συνεισφορές, αυτό, αυτό είναι γνωστό δημοσιεύτηκε και θα δείτε ότι υπάρχουν εκεί πολύ μεγάλοι ρηπαντέ, πολλές μεγάλες χώρες που το έπραξαν ήδη και άλλε ακολουθούν, θα το δείτε των επόμενε εβδομάδε. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Σουηδό Βουλευτή η ευκαιρία αυτή να παρουσιαστεί προ τα έξω με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή, όλοι ω τώρα μιλούσαν για τον πανικό, για τα προβλήματα, τι αρνητικέ πτυχέ. Όχι, να παρουσιάσουμε το θέμα με πιο θετικό τρόπο επιτέλους γιατί έχουμε μια τέτοια ευκαιρία μπροστά μας ε, μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την ε, ενέργεια Α, Πρόεδρος, αυτοί συνάδελφοι ξέρω ότι πλησιάζει η ώρα της ψηφοφορίας και προσέρχονται συνεχώς συνάδελφοι όμως ε, λίγη ησυχία στην αίθουσα λίγη ησυχία στην αίθουσα γιατί αυτά που συζητούμε είναι πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα, μας επηρεάζουν και μας αφορούν όλους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Φιγκέρες. Δεν θα με γρηγορήσω. Έχουμε, είπαμε, ε, αυτούς τους στόχους ε, για το 2050. Ναι, ναι. Και είπαμε ότι αυτό είναι παγκόσμια ρύθμιση, αλλά έχουμε διαφοροποίηση μεταξύ αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Άρα 2030, 2050 ε, είναι πάρα πολύ σημαντική στόχη. Δύο και τους δύο να έχουμε κατά νου και το IPCC θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι έχει γίνει για την ουδετερότητα ε, του διοξιδίου του άνθρακα δηλαδή το πώς θα υπολογίσουμε όλα τα αέρια αλλά και θα υπολογίσουμε με την άλλη μεριά το διοξίδιο. Να, πώς θα έχουμε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2070 που είναι εν προκειμένου η ημερομηνία, άλλα δύο θέματα, άλλα δύο, η συμμόρφωση που είναι θέμα της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται. Είναι μια συζήτηση συναρπαστική, ζωντανή, αλλά πρόκειται να ευθύνονται οι κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν, αλλά και έχουν αρμοδιότητα ελεγκτική και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επίσης, για τον ρόλο αυτών των μη κυβερνητικών ε, φορέων. Πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος που έχουν. Πολλές χώρες δεν ήταν πάρα πολύ εύκολες να το δεχθούν, αλλά τελευταίους 8-12 μήνες υπάρχει κάποιο είδους όθηση προς ε, την κατεύθυνση την επιθυμητή και ελπίζουμε έτσι να τα καταφέρουμε στο Παρίσι. Thank you Πρόεδρος. Κύριε Φιγέρ, σας ευχαριστούμε πολύ. Εξ όλων στην Επιτροπή μας, καλή επιτυχία για τις διαπραγματεύσεις. Συγχαρητήρια επίσης που απαντήσατε όλες τις ερωτήσεις και που τηρήσατε και το χρονικό όριο αυτών των 11 λεπτών που είναι πολύ εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε και καλή τύχη. Δύο λεπτάκια διάλειμμα πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Σε δύο λεπτάκια αρχίζουμε την ψηφοφορία. Okay, dear colleagues, we start the voting. Με uh, Με ψηφοφορίες, συνάδελφοι. Το πρώτο θέμα είναι 106, άρθρο 106, παράταση της περίοδου για το λιφοζέιντ. Για το λιφοζέιντ. Και τώρα είπαμε ότι μπορεί να κάνετε μια δήλωση κύριε Χερμπάντη, ε, όχι παραμονικό με 24 Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου όμω, γιατί θα ήθελα να σα τονίσω πω η Άλντε θεωρείται, θεωρείται ότι έχει πάρα πολύ στριμωχτεί από αυτέ τι ουσίε, γιατί είχαμε θεωρήσει ότι θα εκπνεύσει σχετική περίοδο, όπω είχε πει η Επιτροπή τελευταία του Επομένω, πάσα καθυστέρηση είναι αχώνευτη όμω οποιαδήποτε απόφαση για το να παραταθούν οι χρήσει αυτέ, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση. Αυτό είναι κλασική περίπτωση διεξόδου. Οπότε εμεί ε, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε την Επιτροπή σε αυτό το εξάμεινο το οποίο ζητεί. Ο όμω παραπάνω παράταση δεν θα δεχτούμε. Ευχαριστούμε κύριε Χερμπάντη. Και τώρα για την ΚΟΕ. Κυρία Κονιέτσα. Ευχαριστώ πολύ Επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω να σας παρουσιάσω το αίτημά μας να υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Πολλοί συνάδελφοι δεν ήταν παρόντες για να υπογράψουν το κείμενο, άρα θα ήταν δίκαιο πιστεύω και σωστό για ένα τόσο σημαντικό θέμα να μπορέσουμε να δούμε τι στήριξη υπάρχει ούτω ώστε όλοι να δείξουν την άποψή τους. Να μην κρυφτούν πίσω από την ε, άποψη της, της πολιτικής ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται ένα τέταρτο των μελών της Επιτροπής για να συμφωνηθεί η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα εάν στηρίζεται το αίτημα της Γκουε για ονομαστική ψηφοφορία. Όσοι το στηρίζουν, παρακαλώ να ψηφίσουν ναι. Okay, everybody. όλοι. Πέρας. Ναι, πάνω από το 1 τέταρτο των μελών της Επιτροπής στηρίζουν το αίτημα αυτό. Άρα θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα της ουσίας γλυφοσάτ. Ψηφίζουμε το ίδιο το σχέδιο ψηφίσματος και πάλι ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Everybody has voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Όρια κομπών και έκριση τύπου για κινητήρες εσωτερική καύσης που προορίζεται για μη οδικά κινητά μηχανήματα. Αν αρχίσουμε την ψηφοφορία. Η τροπολογία 68 πρέπει να σε ενημερώσω. Περιέχει ένα λάθος στον κατάλογο ψηφοφοριών λέγεται ότι αν περάσει η συμβαστική 3 τότε καταπίπτει 68 αυτό είναι λάθος ακόμη και αν εγκριθεί λοιπόν η συμβαστική 3 πρέπει να ψηφίσουμε και επί της 68 ωραία ας αρχίσουμε άρθρο 1 τροπολογία 80 του κυρίου ΕΚ Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 81 είναι γλωσσική, δεν την ψηφίζουμε. 82. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ίδιος συσχετισμός. 84 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 Α, έχει αποσυρθεί. Ωραία. 90, 90. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 92. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 μαζί με την 91 ταυτόσημες υπέρ παρακαλώ. Α, καταπίπτουν. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Μαθαίνω, μαθαίνω. 39, συγγνώμη, 93 και 94, με συγχωρείτε, ταυτόσιμες, θα βελτιωθώ. Σας το υπόσχομαι. 93 και 94. Ταυτόσιμες παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 95 υπέρ. Απορρίφθηκε η προηγούμενη. Κατά παρακαλώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι και ΙΜΚΟ εννέα. Ταυτόσημες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 96 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία επί της 96 πέρασε απορρίπτεται 97 και 98 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 99 έχει αποσυρθεί 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καλά έλεγχος άρχεται ελέγχουμε την 102 πέρας oh. Α, είχε έννοια ο έλεγχος. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 100. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάλι με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα και 110. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήμκο 15 υπέρ κατά Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά. Ίμκο 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και εδώ. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο 16. Υπέρ. Η τροπολογία 115 απερίφθη, άρα θα πρέπει τώρα να κρίνουμε την, την ΙΜΚΟ 16 πίνε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά Α, αποχές ας γίνει η ηλεκτρονική ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται Ήμικο 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε για το 118. Πέρας. Απορρίπτω. Συμβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Είναι το 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 σηκώστε το χέρι σας για να είναι ξεκάθαρο ποιος ψηφίζει τι. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά, αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρα Απορρίπτεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα έλεγχο. Ας ελέγξουμε 127. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. 128. Οικονομικός έλεγχος. Πέρας. Απ, απορρίπτεται. 29. Και ταυτόσημη ήμικο 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καλά, ας ελέγξουμε. 130. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Ναι, είχατε δίκιο. Γιατί απορρίπτεται. 131 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 132. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτωται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. 134. 135. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 ε, ψηφίζουμε την ΙΜΚΟ 20, πίνε υπέρ, πίνε κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Αλλά αν θέλετε, ας γίνει παρήθευση για την ΙΜΚΟ 20 ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε, πέρας, απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 15 ε, υπέρ κατά ψηφίζουμε το 15 λέει ο πρόεδρος ή 14 ενεκρίθη Άρα πάμε στο 15. Οπότε και πάλι ψηφίζουμε και πάλι το 15. Είναι υπέρ, είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 21 της ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149. 141 με 152, 137 και 138 157, 149-157 λοιπόν όλες μαζί. Ποιοι υπέρ, ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 και μαζί η ΙΜΚΟ 23 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 24 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. για το 24 της ΙΜΚΟ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. ΥΜΚΟ 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος. ΥΜΚΟ 25 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. ΥΜΚΟ 8 όχι. Όχι καταπληκτή. 163 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός ελέγχος 163 ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. 164 υπέρ και 165 είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 20 26 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 21 και ΙΜΚΟ 27. Όχι, λάθος λέει ο 21 μόνο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ή 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 166 ψηφίσουμε. Πέρας απορρίφθηκαν. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 167 ψηφίζουμε για την 167 πέρας Αφού πιο σημαντική στιγμή. Ήρθε ο Πρόεδρός μας. Εκατόν υπέρ κατά αποχές απορρίβεται ηλεκτρονικός έλεγχος 168 ψηφίζουμε Πέρας. Στο ΕΛΚ είναι ένας παραπάνω. Πέρας της ψηφορίας. Απορρίπτεται. 24 και ήμικο 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 25 του εισηγητή και το 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ, 103 και 104, τρεις από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμικο 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 171 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται Ήμικο 33. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 και Ήμικο 34. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 27 υπέρ μαζί με την 173 και την ήμικο 35 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 και 175 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. ΙΜΚΟ 36 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την ΙΜΚΟ 36 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται Αν θέλετε, ελάτε εδώ. λέω ο πρόεδρος να τα βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, 10 συμβαστικοί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. και ΙΜΚΟ 38 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. καταπίπτει 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 192 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές. Πιστεύω ότι εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. Την 195 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 196 και 197 και 198 unblock μαζί ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απολύπτονται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. απολύπτονται. 200. 201, 205 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απολύτωνε. 202, 203, 204 και ΙΜΚΟ 39 Καυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται πιστεύω νομίζω ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 202, 3, 4 και ΙΜΚΟ 39 ψηφίζουμε Πέρας. Απορρίπτονται. 206, 7 και 8 και ήμικο 40. Μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Τροπολογία 30 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια να βλέπω. κατά. Αποχές. Ε, έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός γιατί είναι 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν ε, σηκώνεται καλά τα χέρια και πού να δω. Αφήστε που κάποιοι άλλαξαν και γνώμη μεταξύ. Στο άρθρο 57 έχω μια προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε την ε, προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβεστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός πιστεύω ότι απορρίπτεται. γιατί 14 συμβαστικοί ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Καλό είναι πάντα να ελέγχει κανείς. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. η ίδια ακριβώ πλειοψηφία εγκρίνεται όπως προηγουμένως. Αλλά ας κάνουμε και έναν ηλεκτρονικό έλεγχο για την συμβαστική 15 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.25 υπέρ. Τροπολογία 225. Ωραία θα ήταν να έχουμε 225 συμβαστικές. Λοιπόν, απλή τροπολογία 225. Κυρία Πυρικά είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 225. Υπέρ. Μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτονται. 2.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.30 ψηφίζουμε της κυρίας Κάντενμπαχ πέρας τροπολογία. 2.33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίβεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί συμβαστική 16 ψηφίζουμε. Συμβαστική 16 είπα. Πέρας. Απολύτωται. Επειδή απορρίφθηκε, πρέπει να δούμε τις αλλε άλλες μία προς μία. 2.34 και 2.43 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτονται. 2.30. Όχι. Α, θέλετε έλεγχο. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. Αυτή τη φορά έφτιαχναν τα μάτια μου. Λοιπόν, 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος 41 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά για την συμβαστική 17 θα ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε. πέρας ψηφορίας απορρίπτεται. Είχα δίκιο. Ήταν σαφές από την αρχή. Τροπολογία. Α, άρα πρέπει να τις δούμε τις υπόλοιπες μία προς μία, να ψηφίσουμε 2.30. 2.40 και 2.44. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 κατά αποχές απορρίπτεται 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε ξεχωριστά τώρα για τις ε, 2.37 υπέρ. Α, μπλοκ 2.37, 41 και 66. 2.37 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2.42 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2.43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Α, ηλεκτρονική ψηφοφορία για έλεγχο. Ε, πέρας. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 2.48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 2.47. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.49 και 2.50 και 2.51 και 2.52 53, 54, 55, 56, 2.57. Α, όχι 2.57. Μέχρι τη 2.56. Όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 2.57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 2.57. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.58 και 2.59 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 2.58 και 9 έλεγχος πέρας απορρίπτονται 2.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 264 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 265 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 και 268 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίτονται 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 και 270 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται αιτιολογικές σκέψεις 1 τροπολογίες 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται συγγνώμη. Ήμκο 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 κατά τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 54. Ψηφίζουμε πέρασμα της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Έχουμε τώρα το τρίτο μέρο. Τι είναι υπέρ. Τι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και σε αυτή την περίπτωση. Το 55. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 και ΕΜΚΟ 3 μαζί. Α, όχι μόνο 56 για την θεολογική σκέψη 12α. Αλλά χωριστά από την 3. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Σηκώστε το χέρι σας. Κατά αποχές αν σαφές, ασαφές ας ελέγξουμε την 56 άρχεται πέρα. Απορρίπτεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 57. Πέρας. Απορρίπτεται. Πολύ αμφίροπα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο να διακρίνει το αποτέλεσμα. Συμβαστική δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε γιατί δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά πέρας απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 61 καταπίπτει 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ κατά εποχές έλεγχος άρχεται για την 68 πέρας απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές και πάλι έλεγχος πέρας απορρίπτεται 71 υπέρ κατά Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 4 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ένα και 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική η ψηφοφορία επί της τροποποιηθήσης προτάσεως ηλεκτρονική άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίσουμε, ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τέλος, απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Και πάλι ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. και παρακαλώ τον κύριο Λαβία να αναλάβει την Προεδρία και σε ευχαριστώ για την συνεργασία. Uh, Να αρχίσουμε την ψηφοφορία για την έκθεση Μπέλετ προς την ε, Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία με την συμβαστική παρθυμονένα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Από ηχές συγκρίνεται. Συμβαστική έξι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα την τροπολογία υπορνών ένα του κυρίου Ξύμπα. Τι είναι υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Φιέλνερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Βιβλία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ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 Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57. Φιέλνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γκέρμπραντι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Ποιε συγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. 86 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Εψηφίζονται. Όλοι πέρασε εγκρίνεται. βογέ 91. Πέτερλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Μπάλας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές κλινικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται και τώρα 109 υπέρ κατά εποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Votiamo l'emendamento 145. Chi è favore? 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 ηλεκτρονικός έλεγχος. Il voto Ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Okay. Il voto è chiuso. Πέρα ψηφορίας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 φιέλνερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Ψηφίσατε όλοι, πέρασε ψηφοφορίες και εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές, λιγονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία και εγκρίνεται. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 πότς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Εγκρίθηκε με μια ψηφοδιαφορά 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε είμαστε στην τελική ψηφοφορία όσον αφορά το σύνολο τη γνωμοδοτήσεω όπω τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε τώρα. Il voto è chiuso, avete votato tutti. Εδώ ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και ευχαριστούμε. Εδώ κυρίσουμε το πέρα της συνεδρίασης και πρόκειται για την επίσημη επόμενη συνεδρίαση. Θα ξαναπούμε στις 22 Δεκάτου